Σοσιαλδημοκράτες και το EFDD αιτήματα ορισμού ε, μελών σε επιτροπές και αντιπροσωπείες. Εάν δεν υπάρξουν ε, κάποιες ενστάσεις, τότε θα εγκριθούν ε, οι ορισμοί αυτών των